Τη σύγκληση, της ασφάλειας, η Ευρώπη ως ε, παγκόσμιος παίκτη και η Ευρώπη των κοινών αξιών. Στον πρώτο πυλώνα των συγκλήσεων η Ρουμανική Προεδρία κατέβαλε τεράστιε προσπάθειες για να προωθήσει τις ε, διαπραγματεύσεις που αφορούν στο μελλοντικό πολιετέ ε, δημοσιονικό πλαίσιο 2021-2027 σε πολιτικό πλάνο αλλά και σε κλαδικό επίπεδο. Κατορθώσαμε επίσης να οριστικοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις σε αρκετά ε, νομοθετικές πράξεις ε, στοχεύοντας την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφάλαιων Αγορών και επίσης για την ενιαία αγορά. Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα τα συγκεκριμένα που ε, είχαμε στο, όπως ε, η ε, εσωτερική αγορά σε όλες αυτές τις πτυχές, ενέργεια, κοινωνικές υποθέσεις, η αλλαγή του κλίματος είναι στοιχεία τα οποία θα παραμείνουν σημεία αναφοράς και ήδη έχουν αναλυθεί από τους εταίρους μας του τρίου, Φιλανδία και Κροατία. Ταυτόχρονα προκλήσεις ε, όπως η ψηφιακή ε, και ε, η οι τεχνολογίες ήταν επίσης θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Συνεισφέραμε στην ενιαία ψηφική αγορά μέσα από την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού. είχαμε πάντα κατά νου τα συμφέρον του πολίτη η ενοποίηση της κοινωνικής πτυχής ε, αντιπροσώπευε μια προτεραιότητα και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Εργασία είναι ένα παράδειγμα επιτυχίας. Από πλευράς Ενεργειακής Ένωσης υιοθετήσαμε την αλλαγή της ε, οδηγίας για το φυσικό αέριο που θα αποτελέσει ένα πλαίσιο ε, ρυθμιστικό διαφανές σχετικά με τις διασυνδέσεις σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο με τρίτα ε, κράτη-μέλη. Παρακολουθήσαμε την ε, ε, ανάπτυξη μια, ενός κοινού οράματος μακροχρόνια ε, προς την ουδετερότητα από πλευρά κλίματος. Ε, εγκρίναμε τις, τους πρώτους κανονισμούς σε ό,τι αφορά τις εκπομπές των βαρέων οχημάτων. Η Ευρώπη της ασφάλειας, ο δεύτερος πυλώνας, ήταν το πλαίσιο στο οποίο δράσαμε για να αυξήσουμε το επίπεδο ασφάλειας, ασφάλειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας κατά νου τις απαιτήσει και τις προσδοκίες των πολιτών. Ολοκληρώσαμε την θητεία της, του φορέα του Οργανισμού Τσακτοφυλακής και Συνεωριοφυλακής μέσα από τη διαλειτουργικότητα. Ε, στέλνουμε έτσι ένα μήνυμα ότι τα συστήματα πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συμπληρωθούν με αμοιβαιότητα. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την συνέχιση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να ερδεωθεί η εσωτερική ασφάλεια και η λειτουργία του χώρου Σέγγεν, ένα στόχο στον οποίο η η Ρουμανία θα ήθελε να συμμετέχει πλήρως στη συνέχεια. Στον τομέα της μετανάστευσης καταβάλαμε προσπάθειες για να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης. Και υπό τις ε, συνθήκες διαφορετικότητας ε, προχωρήσαμε τις διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις για ε, ε, ορισμένες ε, προσωρινές δεσμεύσεις και οριστικοποιήσαμε τις διαπραγματεύσεις για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, των συνδέσμων ε, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά την βελτίωση των αντιδράσεων στις ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έγιναν κάποιες κυρώσεις σε αυτό τον τομέα. Έτσι, για πρώτη φορά θα επιβληθούν κυρώσεις σε άτομα που προσδιορίζονται σε αυτές τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που αποτελούν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη. Η Ρουμανία θα συνεχίσει να δρά σε αυτόν τον χώρο παρακολουθώντας στο στόχο για να ε, φιλοξενήσει έναν ειδικευμένο φορέα σε αυτό το θέμα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πτυχή της δράσης μας ε, στον ε, πυλώνα Ευρώπη παγκόσμιος παίκτης, κάναμε συνεχείς προσπάθειες για να εδραιώσουμε το προφίλ μιας δραστήριας και αποτελεσματικής ένωσης που να εμπλέκεται στη γειτονία της και αξιόπιστης με τις δεσμεύσεις της. Έγιναν πρόοδοι σε σημαντικούς τομείς όπως η περιφέρεια των Δυτικών Βαλκανίων, η εταιρική σχέση με προς και οι σχέσεις με την Μαύρη Θάλασσα. Ε, θέλουμε μια γεωστρατική ε, σχέση για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Δυτικά Βαλκάνια καταφέραμε ε, σε ένα δύσκολο πλαίσιο να διατηρήσουμε τις εξελίξεις της αξιοσημείωτες και τις ιστορικές που έγιναν πέρσι και να διατηρήσουμε τις στρατηγικές ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για τους εταίρους μας στην περιφέρεια και αναφέρομαι στην Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Η συνάφεια των στόχων μας είναι σημαντική στον πυλώνα της Ευρώπης των κοινών αξιών. Το ε, φαινόμενο της παραπληροφόρησης είναι επίκαιρο και Γι' αυτό μεταφέραμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τη διασφάλιση ε, ορθών ευρωπαϊκών εκλογών. Ένας άλλος κύριος στόχος της Προεδρίας μας ε, στόχευε την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της ξενοφοβίας ε, και της ρητορική του μίσους και όλων των μορφών μισαδοδοξίας. Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν από τους εταίρους μας του τρίου. Πιστεύουμε ότι η πρόθεση της ισότητας ευκαιριών και φύλου είναι ένα σημαντικός στόχος που ε, τον ξαναβλέπουμε στην αρχιτεκτονική των νέων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Αναλάβαμε ότι θα δράσουμε για την εδραίωση του ευρωπαϊκού οράματος και ε, κατά το εξάμεινο της Προεδρίας μας καταδείξαμε ότι ε, θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε συνεχείς δράσεις φιλικές προς την Ευρώπη. Ενεπλάκη προσωπικά για την καλή διεκπαιρέωση αυτής της Προεδρίας και από δική μου ε, αποφασιστικότητα ε, λόγω της προσήλωσής μου στο ευρωπαϊκό όραμα. Ανήκω στην γενιά που ορίμασε με αυτή την προσδοκία πλήρως για την ενοποίηση της Ευρώπης και για την αναγνώριση αυτού του θέματος για τη Ρουμανία. Αυτό το αίσθημα ε, της αναγνώρισης της σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες πρέπει να καλλιεργηθεί συνεχώς μέσα από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το όραμα μας δεν πρέπει να προωθεί μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων ούτε ομόκεντρων κύκλων. Η Ρουμανία θα συνεχίσει να προωθεί τον κοινό στόχο εδραίωση του ευρωπαϊκού οράματο και θα παρακολουθεί ταυτόχρονα την οριστικοποίηση της ενοποίησής της. Και αναφέρομαι εδώ σίγουρα στην, ενοποίηση, την πλήρη ενοποίηση στο χώρο Σέγγεν της Ρουμανίας, στο οποίο δρούμε ως de facto μέλος. Θα συνεχίσουμε να δρούμε με πραγματιστικό τρόπο για να ε, προωθήσουμε τις αρχές της δήλωσης του Συμπίου και παραμένουμε προσιλωμένοι στις προσδικίες των δημοκρατικών αρχών και του τους δικαίου. Είναι σημαντικό όμως να μην υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, να μην υπάρχουν χάσματα που να δημιουργούν ε, δύο ταχύτητες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Με την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία επιβεβαίωσε την υπόσταση Ενό πλήρου μέλου που μας δείχνει την ομιμότητα της προσδοκίας μας να ε, κλείσουμε έναν μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευση. Πιστεύω στεναρά ότι το μέλλον μας, όλων μας, δεν μπορεί να το φανταστούμε αλλιώ παρά μόνο στο πλαίσιο μιας πιο ισχυρής, πιο συνεκτικής Ευρώπης προς όφελο τη οποία δουλέψαμε με ενθουσιασμό και επαγγελματισμό και πίστη του τελευταίους έξι μήνες. Έχω την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες της Ρουμανική Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης αντιπροσωπεύουν μία σταθερή βάση για τη συνέχιση της προώθησης ε, της ε, ε, ατζέντα της Ευρώπης την επόμενη περίοδο και εύχομαι στην Φιλανδική Προεδρία κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την στήριξή σας σε αυτό το ε, τελευταίο εξάμεινο για την πολύ καλή συνεργασία και είμαι πεπισμένη ότι η Προεδρία ε, της Ρουμανίας ε, αυτό το τελευταίο εξάμεινο θα παραμείνει στη μνήμη και της Ρουμανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια Προεδρία επιτυχίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ Νταντσίλα και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σεύτσοβιτς, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία ε, Πρωθυπουργέ, αγαπητή Βιορίκα, ε, είναι πάντα μεγάλη χαρά ε, που βρίσκομαι μεταξύ ημών στο Κοινοβούλιο. Σήμερα το πρωί ε, συζητήσατε μάλιστα και τις προσδοκίες και τις κοινές, τα κοινά οράματα για τα επόμενα πέντε χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκινάει και η νέα νομοθετική περίοδος η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα παρουσιάζει πολλές προκλήσεις όπως και πολλές Ευκαιρίε ε, Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο με υψηλές, ε, ισχυρα, ισχυρές εντολές λόγω της μεγάλη συμμετοχή ε, θα ξεκινήσουν μια κοινή πορεία υπέρ της Ευρώπης γιατί εάν θέλουμε να επιτύχει η Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε από κοινού ασκώντας την ευρωπαϊκή τέχνη των συμβιβασμών. Ε, η, τη Ρουμανική Προεδρία μελετούμε σήμερα τον απολογισμό της αλλά βεβαίως και το πνεύμα της εργασίας μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα ήθελα αγαπητή Πρωθυπουργέ, αγαπητή Βιορίκα να σε ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κατέβαλε η ε, Ρουμανία έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμα λίγο πιο, ε, πιο μπροστά την Ευρώπη. Η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, οι χώρες θα πρέπει να δουλέψουν από κοινού ε, και αυτό αποδεικνύεται ε, γιατί 354 προτάσεις που ξεκίνησαν από την ε, Κομισιόν έχουν εγκριθεί οι περισσότερες δε ομοφόνος. Αυτό σημαίνει σκληρή δουλειά και τέχνη του συμβιβασμού και οπωσδήποτε επικοδομητική προσέγγιση. Κατά την έννοια αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρουμανική Προεδρία, ε, τον Πρόεδρο Ιωάννης, ε, την Πρωθυπουργό Νταντσίλα, καθώς επίσης ε, και τους Υπουργούς, χωρίς να ξεχνώ βεβαίως και τον Πρέσβη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους ευχαριστήσω, λίγο, να ευχαριστήσω για τις πολλές επιτυχίες τους. Ε, τον Απρίλιο στην τελευταία ε, Ολομέλεια ε, πραγματικά καταφέρατε να ολοκληρώσετε 95 ψηφίσματα σε, στους πρώτες 100 μέρες της Προεδρία σας. Επίσης το θέμα της ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής είναι ένα, ήταν ένα ιδιαίτερο θέμα, δύσκολο ε, για να το ολοκληρώσετε. Ε, απ' την άλλη πλευρά βέβαια είμαι πολύ ε, ευτυχής γιατί και ο συνάδελφός μου, ο Επίτροπος Αρίας Κανιέτε, είναι εδώ για να σας ευχαριστήσει και αυτός για τα όσα επιτύχατε. Το κοινωνικό θεματολόγιο εξ αρχής ήταν από τις προτεραιότητες ε, της ε, Προεδρίας. Αυτή τη στιγμή ε, ευτυχώς έχει αυξηθεί η δυνατότητα των ανδρών να υποστηρίξουν περισσότερο στη, τις οικογένειες και να υποστηρίξουν ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ πιο εύκολο να προβλέψει κανείς την απασχόληση ακόμα και σε άτυπες μορφές εργασίας. Επίσης, η ε, Ρουμανική Προεδρία, ε, η αρχή για την επιθεώρηση της εργασίας ε, έγινε δυνατότητα. Εξαιρετική εργασία επίσης έγινε και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Μεγάλη πρόοδος έγινε ε, κυρίως σε ε, ένα πολύ κρίσιμο θέμα που είναι το δημοσιονομικό εργαλείο της ε, Ευρωζώνης, θέματα τα οποία θα βρει η επόμενη Προεδρία μπροστά της. Όλα, όλες οι διαπραγματεύσεις, οι δημοσιονομικές, γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Ωστόσο, όταν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να παραχθεί αποτέλεσμα το οποίο να αποτελεί σταθεροποίηση για το μέλλον. Η Ρουμανία έχει αποδείξει ότι σε αυτήν την δύσκολη χρονιά των θεσμικών αλλαγών ε, η Ευρώπη δεν έχει πλέον αυτές, αυτούς τους διαχωρισμούς ε, ε, βορράς, νότος, δύση, ανατολή. Και αυτό φάνηκε την 9η Μαΐου στην διάσκεψη του Σύμπιου. Η τελική δήλωση του ΣΥΜΠΙΟΥ από, τις, ε, από τους 27 ε, ηγέτες ε, κρατών και κυβερνήσεων είναι απόδειξη αυτών που λέγω. Ε, νομίζω ότι, τελειώνοντας πρέπει να πω ότι η Ρουμανία ναι θα πρέπει να γίνει πλήρες μέλος ε, της ε, Σέγγεν και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά το κράτος δικαίου και όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό το ζητούν άλλωστε και οι ίδιοι οι πολίτες. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια πιο σε πιο προσωπικό τόνο ε, πριν ε, και μετά τις ε, μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του κόσμου στην οποία ζούμε πραγματικά μπορούμε να δούμε πόσο άλλαξαν οι χώρες νομίζω και πόσο άλλαξε και η δικιά σας χώρα κάνατε πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι οι πολίτες σας μπορούν και πρέπει να είναι περήφανοι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες εκ μέρου του Λαϊκού Κόμματος. Θα λάβει το λόγο ο κύριος Κόπατσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον πρόεδρο Γιωχάνες, εσάς κυρία Πρωθυπουργέ, του υπουργούς σας και όλους εκείνους που βοήθησαν στο να στεφτεί η πρώτη σας προεδρία από επιτυχία. Αναλάβατε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συζητήσεις που αφορούν ε, στην ανανέωση της Ευρώπης και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Με βάση όλα αυτά είχατε να αντιμετωπίσετε υψηλέ προσδοκίες σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά έπρεπε να δώσει και κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε πρόοδο σε σημαντικά θέματα όπως ε, ψηφιακή αγορά, οδηγία για το αέριο και τραπεζική ένωση. Ο Επίτροπος ήδη αναφέρθηκε σε ορισμένα εξ αυτών. Από κοινού επιτύχαμε επίσης ισχυρή δέσμευση σε ενωσιακό επίπεδο για τη διεύρυνση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Θέλουμε η Προεδρία να διατηρήσει αυτό το σημαντικό θέμα στην ε, ατζέντα της. Ε, η συνάντηση Κορυφή της Σόφιας πρόσφερε ε, τον χάρτη πορείας που είναι απαραίτητος για το ευρωπαϊκό μέλλον αυτής της περιοχής. Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα ε, τις προσπάθειες της Αυστριακής και της Ρουμανικής Προεδρίας στο να προάγουν, να ενισχύσουν αυτά τα κίνητρα. Τώρα πρέπει να δούμε λιγάκι την πραγματικότητα. Αν αποδυναμωθεί αυτός ο δυναμισμός ε, θα υπάρξουν αρνητικές αντιδράσεις ε, και επιπτώσεις στην περιοχή και τρίτες χώρες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή μια κατάσταση που δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανική Προεδρία ξεκίνησε με το σύνθημα συνοχή, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία. Και πράγματι, μια πιο συνεκτική Ευρώπη είναι μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Έκλεισαν επιτυχημένα πολλά σημαντικά χαρτοφυλάκια και θέλω να επισημάνω κυρίως ε, τη συμφωνία για τη ρύθμιση των ευρωπαϊκών συνόρων και της ακτοφυλακής. Το να ενισχύσουμε εκεί τις δυνατότητές μας, αυτό ανέκαθεν ήταν προτεραιότητα για μας. Η πιο σημαντική ε, ε, ελευθερία των πολιτών μας είναι το ότι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να τη διασφαλίσουμε αυτή την ελευθερία μόνο αν ε, φυλάσσουμε καλά τα εξωτερικά μας σύνορα. Όσον αφορά τη χώρα μου, τη Βουλγαρία, νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ καλό παράδειγμα ως προς την εξασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων. Εκεί μας έχει βοηθήσει βέβαια και η ελεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα του ΕΛΚΑ είναι υπέρ του να υπάρχουν πιο ισχυρά ευρωπαϊκά σύνορα, να υπάρχει ευρωπαϊκή ακτοφυλακή που να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς καθυστέρηση μόλις μια χώρα αντιμετωπίσει μεταναστευτικές πιέσεις. Στηρίζουμε την ενίσχυση της Frontex με 10.000 νέους σύνοριοφύλακες. Ένα άλλο βασικό θέμα ήταν η συζήτηση για το σε δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο. Το ΕΛ καθέλει μια φιλόδοξη Ευρώπη Χρειαζόμαστε τα μέσα για να μπορούμε να ε, επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις επιθυμίες των πολιτών της αν δεν έχει και τα απαραίτητα μέσα. Ε, θέλουμε βέβαια οι διαπραγματεύσει να θέλαμε να ολοκληρωθούν πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά παρόλα αυτά συγχαίρουμε τη Ρωμανική Προεδρία για αυτά που πέτυχε. Είναι σημαντικό να μην μειώσουμε τους πόρους από τον προεπλογισμό που διοχετεύονται στην ε, πολιτική συνοχής. Ε, τα ε, επενδυτικά ταμεία βοηθούν στο να μειωθεί το χάσμα και αντιμετωπίζουν και την φτώχεια. Όλοι μας λοιπόν πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι ε, συγχαίρουμε τη Ρουμανική Προεδρία και για τις συζητήσεις σχετικά ε, με τις σχέσεις καλής γειτονίας, κυρίως προς ε, ανατολικά. Δυστυχώς βέβαια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ακόμα δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν. Συνεχίσατε τις ε, διαπραγματεύσεις για τον διορισμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Εμείς στηρίζουμε τις ε, προσπάθειές σας για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Βεβαίως η Ένωσή μας δεν είναι μόνο οικονομική, ε, δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίζουν ρόλο, ρόλο παίζουν και οι αξίες. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κράτος δικαίου είναι μια θεμελιώδης αξία που ενδιαφέρει εμάς ε, το ΕΛΚ. Και τέλος, όσον αφορά το ρόλο της Προεδρίας, η Προεδρία έχει ως μέλημα να καθορίσει και στρατηγικές προτεραιότητες για το μέλλον. Και εδώ μια σημαντική επιτυχία είναι η συνάντηση κορυφής που οργανώθηκε στο Σύμπιο από τον πρόεδρο Ιωάννης. Εκεί υπογράφηκε η δήλωση του Σύμπιου ένα βήμα προς μια πιο ισχυρή δημοκρατική ένωση. Λάβαμε ισχυρή εντολή από τους πολίτες μας. Πάνω από 50% των πολιτών μας πήγαν στις ευρωπαϊκές εκλογές και τώρα είναι η σειρά της Φινλανδικής Προεδρίας να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Ελπίζουμε, Πρόεδρος, θα εκλεγεί σήμερα το απόγευμα ε, η κυρία Φόντερ και θέλουμε μαζί να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο πρόγραμμα που μας παρουσίασε σήμερα το πρωί η υποψήφια Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειές σας και προσβλέπουμε στην Φινλανδική Προεδρία. Η κυρία Γκαρσία Πέρες, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Πρωθυπουργέ, η Ρουμανία να ε, ίσκησε την Προεδρία ε, κατά μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και λόγω του Brexit αλλά ε, και λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που είχατε για να εργαστείτε και λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών. Ωστόσο αυτοί οι μήνες ήταν πραγματικά καρποφόροι και θα ήθελα να συγχαρώ την Ρουμανία και να καλωσορίσω στην Ολομέλεια την την Πρωθυπουργό της ε, χώρας, κυρία Νταντσίλα Βιορίκα. Έγινε σημαντική δουλειά προετοιμασίας ε, του εδάφους για μια ενδεχόμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου που θα είχε όσο γίνεται λιγότερη επίπτωση και για τους Βρετανούς πολίτες αλλά και για τους υπόλοιπους ε, πολίτες. Αυτό κάνατε εσείς στη διάρκεια της Προεδρίας, να δίνετε απαντήσεις στους προβληματισμούς των πολιτών με τον τρόπο τρόπο αυτό ε, δείξατε και αλληλεγγύη, αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλές οι περιφέρειες που απεριμόνονται, διότι οι νέοι δεν βλέπουν ε, μέλλον σε αυτές. Το, ε, το θέμα της συνοχής οπωσδήποτε ήρξε πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως όλοι οι πολίτες να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες έτσι, και αυτό να γίνει υπέρ και των ε, περιφερειών. Ε, πολλά σημαντικά κείμενα ε, περάσατε. Μεταξύ αυτών θα ήθελα να αναφερθώ στην προπαρασκευαστική εργασία και τις συμφωνίες όσον αφορά το ΠΔΠ για τα επόμενα 7 χρόνια. Αυτός ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι απαραίτητος για την θητεία που ξεκινάει τώρα. Μονάχα με ισχυρό λέω προπολογισμό θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πολιτικέ που χρειάζονται όλοι οι πολίτε και όλες οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγαλύτερη προστασία επίσης των ε, εργαζομένων μέσα από ένα κείμενο το οποίο αφορά ακριβώς τις δικαιότερες προϋποθέσεις ε, εργασίας. Και αυτό ήταν θεμελιώδος σημασία για μας. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω ως μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης θητείας ήταν ε, η, αυτή η οποία αφορούσε τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ε, μέσω της οποίας προβλέπεται για πρώτη φορά η πατρική άδεια. Επίσης ε, σε θέματα ε, ισότητας φύλων, ισότητας ευκαιριών, τα πρόθεσε τα θέματα αυτά η Ρουμανική Προεδρία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας συγχαρώ και για τις, ε, κυρίως για τις πρωτοβουλίες που πήρατε ε, κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αγαπητή κυρία Νταντσίλα, αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, θα δώσετε τώρα τη σκητάλη σε μια νέα ε, προεδρία έτσι ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη πιο σωστή και πιο δίκαιη αυτό που ζητούν και οι πολίτες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, από την ομάδα Renew Europe ο κύριο Τουντοράτσε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ Ταντσίλα, Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Σεύκοβιτς, η πρώτη Προεδρία της Ρουμανίας ήταν μια ε, Προεδρία των Αντιθέσεων σε τεχνικό επίπεδο, οι διπλωμάτες και οι τεχνοκράτες κατάρθωσαν να κλείσουν 90 ε, θέματα. Θα ήθελα να συγχαρώ τους επαγγελματίε πίσω από τη σκηνή που πολύ σπάνια τους ευχαριστούμε για το έργο που επιτέλεσαν για την επιτυχία αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια και το πολιτικό επίπεδο αυτής της Προέδριας. Ε, λυπάμαι να πω ότι η σημερινή κυβέρνηση της Ρουμανίας απασχολήθηκε ε, πολύ περισσότερο με τα θέματα της δικαιοσύνης ε, στη χώρα τους. Αυτή, εδώ είχαμε και μια ρητορική αντιευρωπαϊκή και λαϊκιστική. Ευτυχώς σε αυτή τη ρητορική ε, τιμωρήθηκε από τους Ρουμάνους στη ψηφοφορία. Η Ρουμανία δείξε ότι είναι περισσότερο παρά η πολιτική που αντιπροσωπεύει. Η Ρουμανία σημαίνει πρώτα απ' όλα πολίτε που κάθισαν στι ουρέ για να ψηφίσουν για τι εκλογέ. Ε, άξιζαν περισσότερα για αυτέ τι ευκαιρίε που έρχεται μία φορά κάθε 14 χρόνια. Μετά από αυτή την Προεδρία, ε, έχουμε πολλά θέματα τα οποία δεν κατορθώσαμε να προωθήσουμε τους τελευταίους μήνες. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία τέτοια θέματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ε, το θέμα του PDP. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το προηγούμενο η Δελταπή οδήγησε σε ακύρωση κάποιων θεμάτων. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε επαρκεί πόρου για την αγροτική πολιτική και μια πολιτική συνοχής που να διασφαλίζει την πραγματική σύγκληση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στο θέμα της παιδείας και της υγείας ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων για ελάχιστα επίπεδα ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, χρειάζεται να ε, ξεμπλοκάρουμε ε, το ε, θέμα του ε, Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Θα πρέπει να γίνει ε, άμεσα αυτό το πράγμα. Αναμένω από την Φιλανδική Προεδρία να έρθει την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε αυτό το θέμα. Τρίτον, πρέπει να προωθήσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση και την διαχείριση των συνόρων. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος για το χώρο του Σέγγεν, για το μέλλον του χώρου του Σέγγεν, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα κράτος μέλος πίσω και να μην αμφισβητείται πια ε, η διαδικασία αυτή για κάποιες χώρες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Λαμπέρ, εξ ονόματος των Πρασίνων, 3,5 λεπτά. Καλώς ορίσατε, κυρία Πρωθυπουργέ. Χαιρόμαστε πάντα όταν εδώ στην Ολομέλεια υποδεχόμαστε ε, έναν αρχηγό ε, κράτους. Ε, εντάξει, ε, ε, καμιά φορά λέμε ότι το Συμβούλιο δεν έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση αλλά είστε νομιμοποιημένοι ε, στις ε, ε, χώρες σας και έχετε την ευκαιρία όταν έχετε την Προεδρία να δείξετε τι μπορείτε να κάνετε και είναι γεγονός ότι η Ρουμανική Προεδρία πραγματικά της βγάζουμε το καπέλο όσον αφορά την διοικητική εργασία. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου και όταν γνωρίζουμε ε, και την πίεση, την τεράστια πίεση για να προωθηθούν ε, κάποιοι φάκελοι, πραγματικά ε, η επιτυχία είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν και κάποια, κάποιοι φάκελοι οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους 90 που όμως είναι εμβληματική σημασία. Το ίδιο το Συμβούλιο σε κάθε μία από τις συνεδριάσεις του κουνάει μπροστά από όλους αυτό το φάκελο για την μετανάστευση και το άσυλο ε, καμονόμενο ότι ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό και κανένα άλλο δεν είναι τόσο σημαντικό εδώ και τέσσερα χρόνια. Αυτό ακούμε. Κάθε φορά στα συμβούλια, κάθε φορά στα συμπεράσματα αυτό ακούμε. Ε, μετανάστευση, μετανάστευση, ξαναμετανάστευση, διαχείριση συνόρων κτλ. Και τελικά περιμένουμε ακόμα μία θέση του Συμβουλίου όσον αφορά αυτή τη δέσμη που έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την μεταρρύθμιση του ασύλου και που δεν βλέπουμε ε, να προχωράει. Τι κάνατε έτσι ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα. Ε, ένας από τους λιγότερο ορατούς ρόλους της Προεδρίας είναι να ξεμπλοκάρει ε, κάποιους φακέλους αποφασίσατε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει ομόφωνα να αποφασίζει ε, και σημαίνει αυτό ότι ένα κράτος μέλος και σας βεβαιώ ότι είναι παραπάνω από ένα τα κράτη-μέλη που θέλουν να μπλοκάρουν μπορούν να το πράξουν. Αλλά ε, πραγματικά δεν κάνετε τίποτα, δεν κουνάτε το μικρό σας δαχτυλάκι. Ε, και ε, τελικά όλοι το ίδιο κάνουν. Κανένας δεν είναι καλύτερος. Ε, ο προλαλή σα επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα της φήμη. Όταν μία χώρα ηγείται της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, αυτή η χώρα κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει, ενσαρκώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. και η κυβέρνησή σας η κυβέρνηση, το τονίζω, όχι η Ουγγαρία, ούτε η Πολωνία, ούτε η Ρουμανία που ε, απολύτως έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που κυβερνούν είναι ε, μια κυβέρνηση η οποία με πάρα πολύ άγριο τρόπο κατέστηλαν ειρηνικέ διαδηλώσεις πριν από ένα χρόνο. Η δικιά σας χώρα, η δικιά σας ε, κυβέρνηση. Ε, πραγματικά πρόκειται για μια ε, περίπτωση πραγματικής αιμονής όσον αφορά αυτά τα θέματα. Και άλλωστε ο κόσμος τη ζητούσε, ζητούσε να καταδικαστούν για διαφθορά η πολιτικοί. Αυτό είναι ε, ε, πολύ δυστυχές και νομίζω ότι και το Συμβούλιο και ε, το όργανο κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτή η ομάδα της Βενετίας πραγματικά μένουν κενό γράμμα στην ουσία γιατί εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενώ από την άλλη μεριά περιμένουμε ακόμα την ακρόασή του και περιμένουμε ακόμα να δούμε καταστάσεις οι οποίες θα τιμούν την Ευρώπη ενώ αυτά που είδαμε δεν τιμούν ούτε την Ευρώπη ούτε τη Ρουμανία. Η Ρουμανία αξίζει καλύτερα και περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Σεμπέ εκ μέρους της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία. Παρακαλώ. Κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρία, επανειλημμένα πήγα στο Βουκουρέστι για τη διάσκεψη των Προέδρων ε, τον Νοέμβριο, αλλά ε, και στη διάσκεψη των μέλων της Ευρώπης. Κάθε φορά εμείς ε, θίξαμε τα, τα μεγάλα διακυβεύματα, τις μεγάλες προκλήσεις που οι πολίτε θα πρέπει σε ολόκληρη την Ευρώπη να αντιμετωπίσουν. Οργάνωση τη οικονομία, προστασία δεδομένων, προστασία των ε, ε, συνόρων, ε, εκβιομηχάνηση και διατήρηση του γεωργικού ιστού. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να είναι ε, όχι αποτελεσματική ούτε καν παρούσα. Όσον αφορά τις ε, ελεύθερες ε, συναλλαγέ. το είδαμε πρόσφατα με το Βιετνάμ και τις χώρες Λατινική Αμερικής, προσπαθεί να γίνεται όσο, όσο γίνεται πιο καταστροφική για ολόκληρο τον πλανήτη. Πρέπει να πούμε για την Ρουμανική Προεδρία ότι οπωσδήποτε αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο και υποχείριο Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, η οποία ε, ε, παίρνει αποφάσεις ενάντια στη βούληση των λαών. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις προτάσεις, ελέγχει τις, την εφαρμογή των κειμένων, αλλά υποτίθεται ότι είναι και ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Οι γραφειοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ε, ε, ε, κυβερνήσουν κατά κάποιο τρόπο την Ευρώπη. Και 38 παράδειγμα είναι ο κύριος Τίμερμαν ο οποίο θα κρατήσει τη θέση του, θα κρατήσει τις αρχές του, έτσι ώστε σιγά σιγά να στραφεί ξανά κατά της Ιταλίας, κατά του Σαλβίνη, προσπαθώντας να αποσυντονίσει και να αποσταθεροποιήσει δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Η Ανατολική Ευρώπη είναι ο μεγάλος λησμονημένος ε, στις ε, ε, θέσεις των επικεφαλής των οργάνων. Στην ουσία η Γερμανία, η καγκελάριος της Γερμανίας, οι αχυράνθρωποι της, οι εκπρόσωποι της είναι αυτοί που παίρνουν παντού τις θέσεις έχοντας ε, υπομείνει το ζυγό του κομμουνισμού, η κεντρική και ανατολική Ευρώπη χρειάζεται ηγέτες δυνατούς έτσι ώστε ε, να αναλυφθούν υποχρεώσεις και όσον αφορά και το θέμα της υποχρεωτικής κατανομής ε, των μεταναστών. Η Επιτροπή Juncker δεν κατάφερε τίποτα. Μπλοκαρίστηκε η μεταρρύθμιση της, του Δουβλίνου κυρίως από την Ουγγαρία και την ε, Πολωνία. Αλλά και οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν έδωσαν την δυνατότητα ε, ε, βέβαια να διευρύνει την θέση κάποιων, την παρουσία κάποιων θέσεων, αλλά τουλάχιστον δεν προχωρήσαμε και πολύ προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι θετικό. Απ' την άλλη πλευρά, η επικεφαλής της Κομισιόν μαζί και με την Προεδρία της Φιλανδίας θα μπορούσε δυστυχώ να οδηγήσει σε μεγαλύτερο φεντεραλισμό, σε περισσότερη ε, ελευθερία, σε περισσότερους μετανάστες που θα μπαίνουν στα σύνορά μα. Ε, και στην ουσία να δημιουργηθεί έτσι μία μηχανή η οποία θα κατατροπώσει την Ευρώπη. Εκ μέρου του ECR, η κυρία παρακαλώ. Η πρώτη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήρθε σε ε, δύσκολες στιγμές όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμαζόταν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και πριν από τις ευρωεκλογέ. Παρά ε, τις χαοτικές ε, περιστάσεις η Ρουμανία απέδειξε ότι ε, ανταποκρίθηκε στους στόχους που ήθελε να πετύχει. Η Ρουμανική Προεδρία θα μείνει στη μνήμη μας για κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες και σημαντικές συμφωνίες όπως είναι η οδηγία για το αέριο, για την ψηφιακή Ευρώπη, πρώτο πρόγραμμα ε, για τους ε, κανόνες για τις εκπομπές ε, ε του άνθρακα για βαρέα οχήματα κλπ. Παρόλο που μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα στον τομέα της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, η Ρουμανική Προεδρία ε, μπορεί να θέσει ως παράδειγμα ότι ακόμη και ε, νέα κράτη-μέλη έχουν ε, σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο να παίξουν Δυστυχώς εκείνοι που υποτίθεται ότι έπρεπε να δουν το ορμανικό παράδειγμα ως ευκαιρία ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση και τα νέα μέλη ε, παρέμειναν αδρανείς ε, και ε, στην επιλογή των νέων ηγετών περιθωριοποιήθηκαν αυτές οι χώρες. Αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν είναι καλό για τους νέους Ευρωπαίους ε, που θέλουν να αναπτυχθούν σε νέα ε, δημοκρατικά ευρωπαϊκά πρότυπα η ε, επιλογή των ηγετών έχει δείξει, παρόλο που ε, η Ιρμανία έδειξε ότι σε αυτή την Ευρώπη υπάρχει φιλοδοξία και γνώση για να συμβάλλουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Ε, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη των νέων δημοκρατιών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των οποίων η ανάπτυξη ακολούθησε διαφορετική διαδρομή, αυτό αυξάνεται όλο ένα. Είναι σαφές ότι τα παλαιότερα μέλη θέλουν να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους φορά που αναλαμβάνονται αποφάσεις. Ε, έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από αυτούς, αλλά ε, η Νέα Ευρώπη δεν πρέπει να παραμείνει ε, υπόδουλο της παλιάς Ευρώπης. Θα θέλαμε να δούμε την Ευρώπη να αξίζει το σύνθημα ενωμένη στη διαφορετικότητα και να σταματήσουμε ε, να θέλουμε συνεχώς την ομοιομορφία και την, τον συγκεντρωτισμό διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές συγκρούσεις που σίγουρα θα είναι καταστροφικές για την Ένωση. Ο κύριος Παπαδημούλης Δημήτρη παρακαλώ από την κούε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Νταντσίλα αλλά και κύριε Σεύκοβιτς συζητάμε τον απολογισμό της Ρουμανικής Προεδρίας περίπου δύο ώρες πριν το ευρωκοινοβούλιο ψηφίσει για τη νέα προτινόμενη πρόεδρο της κομισιόν. η προεδρία σας διεξήχθη ένα δύσκολο εξάμεινο με ευρωεκλογές με το brexit να κινείται από τη μία αβεβαιότητα στην άλλη και με οξυμένα τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. έχετε στο ενεργητικό σας ότι καταφέρατε να κλείσετε αρκετούς φακέλους που εκκρεμούσαν και αυτό καταγράφεται στα θετικά της Ρουμανικής Προεδρίας. Αλλά τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωκοινοβούλιο και απασχολούν και τους πολίτες των κρατών μελών έμειναν σε εκκρεμότητα. Δεν προχώρησαν. Δεν προχώρησε προς τα μπρος η απέτηση των πολιτών για ένα πιο ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό που να στηρίξει και να μην αποδυναμώσει τις πολιτικές συνοχής γιατί οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες ενισχύονται. Δεν προχώρησε ο κοινωνικός πυλώνας ο οποίος παραμένει μια ετικέτα κύριε Σεύκοβιτς μετά τον Γκέτεμποργκ... χωρίς δεσμευτικές πολιτικές που να τον κάνουν πράξη. Δεν έγιναν βήματα για να αρχίσει να συζητείται και επιτέλους να αρχίσει να εφαρμόζεται ένας κατώτατος υποχρεωτικός ευρωπαϊκός μισθός παντού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν λίγες ώρες τον υποσχέθηκε και πάλι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και πριν πέντε χρόνια τον είχα ακούσει από τον κύριο Γιούνκερ και ακόμη είμαστε στο σημείο μηδέν. Επειδή δεν θέλω να είμαι άδικος, θέλω να πω ότι έγιναν και θετικά βήματα όπως η προετοιμασία από το συμβούλιο επί προεδρίας των κυρώσεων εναντίον της επιθετικότητας της τουρκικής ηγεσίας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και είμαι βέβαιος ότι και η φιλανδική προεδρία θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο γιατί οφείλουμε να στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές αξίες όταν απειλούνται από επιθετικές συμπεριφορές γειτόνων της ευρωπαϊκής ένωσης όπως επίσης θεωρώ ότι θετικό ότι προσπαθήσατε στον χώρο της νοτιοανατολικής ευρώπης να συνεχίσετε το θετικό παράδειγμα που άνοιξε η συμφωνία των πρεσπών μεταξύ της πατρίδας μου της ελλάδας και της βόρειας μακεδονίας και εκτιμώ ότι και η νέα κυβέρνηση της ελλάδας σε αντίθεση με όσα έλεγε προεκλογικά θα συνεχίσει να σέβεται και να εφαρμόζει αυτή τη συμφωνία. τελειώνω κυρία νταντσίλα με μια έκκληση στο πρόσωπό σας εξ ονόματος όχι μόνο της πολιτικής μου ομάδας αλλά και πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων και ξέρω ότι και η Κομισιόν συμμερίζεται αυτή την έκκληση. Σας ζητώ να σταματήσετε τώρα την βάρβαρη μεταφορά με άθλιες συνθήκες 70.000 προβάτων από τη Ρουμανία στον Περσικό κόλπο, διότι αυτό παραβιάζει κάθε έννοια πολιτισμού που πρέπει να σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα των ζώων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς από το κόμμα του Brexit ε, θεωρούμε ότι όλοι πιστεύετε ότι κάνουμε τις χειρότερες ομιλίες, τις ε, λιγότερο δημοφιλείς ε, σε αυτήν την αίθουσα, αλλά ο κύριος από τους πράσινους έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη. Ε, προσπάθησε να σας πει τι πρέπει να κάνετε στη χώρα σας. Αξιοσημείωτο. Αλλά ε, όσον αφορά τη Ρουμανική Προεδρία που τελειώνει, που τελείωσε. Θα ήθελα να συγχαρώ κυρίως τη Σιμώνα Χάλα για την ε, πολύ καλή απόδοσή της στο Wimbledon το Σάββατο. Ήταν μια απόδοση δύναμης, ε, ακρίβειας και το ακόμα πιο σημαντικό φαντάζομαι ότι θα ενέπνευσε εκατομμύρια κορίτσια στη Ρουμανία και αλλού για να συμμετάσχουν στον αθλητισμό. Ε, βεβαίως ε, η συλλογική περηφάνεια για την απόδοσή της ε, δείχνει ότι οι Ρουμάνοι νιώθουν περήφανοι. Είναι υπερήφανοι για την ταυτότητά τους. Δεν μιλάω για εθνικισμό, ίσως κάποιοι να ήθελαν να το ακούσουν αυτό, αλλά αυτοί που ήθελαν να το ακούσουν δεν είναι παρόντες. Οι ρουμανικές σημαίες κοιμάτισαν ε, από το Βουκορέστι μέχρι και πολύ πιο απομακρυσμένα μέρη. Δεν ακούστηκε βέβαια ο ενωσιακός ύμνος. Ο αθλητισμός μπορεί να κάνει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο για να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Δυστυχώς, οποτεδήποτε υπάρχουν προθέσεις για ευρωπαϊκά εγχειρήματα, τότε διαπιστώνουμε μεγαλύτερη διαίρεση από ενότητα. Ε, πανέρχομαι στους τέσσερις πυλώνες που αναφέρεται, κυρία Πρωθυπουργέ. Ας ε, κρίνουμε με τις ίδιες ε, προτεραιότητες. Εσείς μιλήσατε για τη σύγκληση μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χαμηλότερη τα τελευταία 30 χρόνια. 16% ενεργεία των νέων, 20% στη Γαλλία, 30% ε, στην Ιταλία και την Ισπανία, 40% στην Ελλάδα. Ολόκληρες γενιές νέων έχουν ε, καταστραφεί ε, δεν πιστεύουν στο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Μετά, όσον αφορά τη δυνατότητα άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το δικό της το στρατό και αυτό ενθαρρύνει όμως εκείνους που θέλουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια της Ευρώπης μέσα από το ΝΑΤΟ. Για όσους από εσάς θα παραμείνουν εδώ όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας πω πολύ σύντομα. Ίσως να περιμένετε περισσότερα από τη Φινλανδική αλλά πιστεύω ότι αυτό θα είναι τρίαμβος ε, της απογοήτευσης υπερβολικών ε, ε, προσδοκιών. Ας εορτάσουμε λοιπόν την επιτυχία της Σιμώνα Χάλεκ, ένα πραγματικό σύμβολο της ρουμανικής υπερηφάνειας που δεν ζημίωσε ούτε την οικονομία ούτε την ασφάλεια στην Ευρώπη. adesso... Και τώρα ο Αντιπρόεδρος ε, κύριος Σεύκοβιτς ε, για να ε, τοποθετηθεί στη δεύτερη παρέμβασή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές ε, για το ότι επισήμαναν τις ε, προκλήσεις ε, που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε οποτεδήποτε προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια κοινή μη διαιρεμένη Ευρώπη και συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο στον κοινωνικό μας πυλώνα και είμαι σίγουρος ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη στο θέμα του κατώτατου μισθού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Όπω ακριβώ πρότεινε η κυρία Γκάρσια Πέρε. Θα ήθελα όμω να ευχαριστήσω και για το ότι επισημάνατε τι επιτυχίε τη Ρουμανική Προεδρία. Ο κύριο Κόπατσιτ το έκανε, ανέφερε όλου του σημαντικού φακέλου που ολοκληρώθηκαν χάρη του επαγγελματισμού των Ευρωπαίων διπλωματών και υπουργών. Επίσης, να επισημάνω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τη Ρουμανική Προεδρία στο να ολοκληρώσουμε ε, φακέλους που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Πολλά λοιπόν έγιναν σε χρόνο ρεκόρ, διότι η Ρουμανική Προεδρία ξεκίνησε ε, σε μια μεταβατική φάση όπου ο χρόνος για πραγματική νομοθετική δουλειά ήταν πολύ περιορισμένος αλλά τον εκμεταλλευτήκατε σωστά και επαγγελματικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά να επισημάνω ότι κατορθώσατε να κάνετε αυτή την πολύ σκληρή δουλειά παρότι ήταν η πρώτη σας προεδρία. Γνωρίζω πολύ καλά ε, πόσο κερδίζει ένα κράτος μέλος από τέτοια εμπειρία, από το να υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις με άλλους εταίρους και άλλους θεσμούς. Άρα δηλαδή ήταν ε, όχι μόνο επένδυση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που μάθατε θα μεταφραστούν σε μεγαλύτερο επαγγελματισμό της διοίκηση στη Ρουμανία. Είμαι σίγουρος ότι όλη αυτή η δουλειά που επενδύθηκε στην Ευρώπη θα σας επιστραφεί ε, και με το παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρώτη σας προεδρία. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεύκοβιτς και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Πρωθυπουργό την κυρία Ντάντσιλα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχαριστίες. Πραγματικά είχαμε την Προεδρία σε μία περίοδο γεμάτη προκλήσεις τις οποίες δεν είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή και αναφέρομαι στη διαδικασία του Brexit, στο γεγονό ότι υπήρχαν οι ευρωεκλογέ, έτσι ώστε όλη η δραστηριότητα της Προεδρίας έπρεπε να συγκεντρωθεί στις πρώτες 100 μέρες. Πραγματικά ε, ε, θα, θέλαμε να κλείσουμε 100 ντοσιέ, κλείσαμε 90, αλλά κάναμε πολλά βήματα μπροστά και πράγματι, κύριε Αντιπρόεδρε, για τη Ρουμανία είναι ένας λόγος για να το γιορτάσουμε. Να το γιορτάσει όλος ο λαός μας, όλοι όσοι πιστεύουν στη Ρουμανία, όλοι όσοι θέλουν να αντιπροσωπεύουν αξιοπρεπώς τη Ρουμανία. Όντως, είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα και το επιθυμούσαμε αυτό αλλά δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις αυτή την συνένεση ανάμεσα σε 28 κράτη-μέλη με διαφορετικές προτεραιότητες το καθένα και ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα πρέπει εμείς να είμαστε ένας πολύ καλός διαμεσολαβητής, διευκολυντής και πιστεύω ότι η Ρουμανία αυτό το πέτυχε και κατάφερε να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα. Σχετικά με το ΠΔΠ, ε, πράγματι είμαι πεπισμένη ότι το νέο κοινοβούλιο ε, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα εξασφαλίσουν αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική προοπτική και τις προβλέψεις, αλλά και σε αυτό το κεφάλαιο κάναμε εμείς ως Προεδρία σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την πολιτική της συνοχής, αλλά και σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Τα έργα μπορούν να συνεχιστούν, αλλά για να έχει την αποτελεσματικότητα που όλοι θέλουμε ένα έργο θα πρέπει να έχει και ε, την χρηματοδοτική προοπτική. Ε, επιλέξαμε την συνοχή διότι πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε συνοχή και ενότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μόνο εάν ε, καταδείξουμε ότι υπάρχει συνοχή μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά και μπορεί να κάνουμε μεγάλα βήματα μαζί. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συνοχή είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας προεδρίας, αλλά η συνοχή θα πρέπει να οδηγεί και να καθοδηγεί τις δράσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικά. Κύριε Τουντοράκε, θα σας απαντήσω ιδιαιτέρως. Ε, οι τεχνοκράτες και οι διπλωμάτες της Ρουμανίας ε, δεν είναι αυτοί που ε, κάναν την Προεδρία. Την Προεδρία καθοδήγησε η κυβέρνηση. Σε κάθε συνάντηση ο, κάποιος υπουργός ήταν επικεφαλής. Υπήρχε μια πολύ αγαστή συνεργασία ανάμεσα σε όλους όσους, όσοι ανεπλάγησαν, όσοι έδρασαν με, πραγματικά για τη Ρουμανία και όχι ενάντια στη Ρουμανία. Πριν από μερικά λεπτά με ρώτησε κάποιο, πιστεύετε ότι οι, Ευρωπαίοι, οι Ρουμάνοι Ευρωβουλευτέ θα ενωθούν για να βελτιώσουν την εικόνα της Ρουμανίας και είπα ναι, τώρα φεύγω απογοητευμένη. Άτομα σαν και εσάς δεν θα δώσουν κάτι θετικό στη Ρουμανία. Αφήστε τα προβλήματα στη χώρα μας. Μην τα φέρνετε στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι αυτά τα πράγματα δεν δίνουν κάτι επιπρόσθετο στην εικόνα της χώρας μας. Επίσης όλοι συγχάρηκαν την Ρουμανική Προεδρία έγιναν ε, ορισμένα πράγματα ε, Πίστευαν κάποιοι ότι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά δεν μας επέκριναν και εδώ δεν θα δείτε πολλούς ευρωβουλευτές που να επικρίνουν τη χώρα τους. Αλλά εσείς το κάνατε ακριβώς όταν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι στη Ουρμανία υπάρχει λόγος να γιορτάζει κανείς. Και ακόμη περισσότερο θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, μάθετε λίγο πριν ε, να μιλάτε, ε, έχει έργα ε, να καταδείξει. Μιλήσατε και για τρία θέματα που δεν γνωρίζετε και πιστεύω ότι δεν ξέρετε τίποτα για τις, ε, τα επιτεύγματα της Ρουμανίας στην Προεδρία της. Δεν ότι δεν ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια μιας Προεδρίας μια χώρα δεν μπορεί να παρέμβει. Πρέπει να είναι διευκολυντής και αυτό ακριβώς έκανε η Ρουμανία και θα χαιρόμουν αν σε αυτό το πολύ σημαντικό ε, έργο για την χώρα μου, το πολύ σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αν υπήρχε συνένεση γιατί έχω βρει την συνένεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω αντιμετωπίσει την συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχω αντιμετωπίσει ε, συνένεση ανάμεσα σε πολλούς ευρωβουλευτές, ε, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλοι αντιληφθήκαμε και καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή και αν δεν δράσουμε ενωμένα δεν θα ε, δώσουμε μια καλή κατεύθυνση στο οικοδόμημα της Ευρώπης και ακούσαμε όλες τις συμβουλές και όλοι μαζί πετύχαμε αυτό που πετύχαμε. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει μας καθοδηγήσει και στην ε, περίοδο που θα ακολουθήσει. Να δώσουμε προστιθέμενη αξία. Οι πολίτες δεν χρειάζονται σκάνδαλα, χρειάζονται πράγματα που να τους βοηθούν στην καθημερινότητά τους. Πιο, πολιτικές πιο κοντά σε αυτούς, όχι πράγματα που να τα βγάζουμε στο δημόσιο χώρο νομίζοντας ότι αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά από πολιτικής άποψης. Κύριε Λάμπερτς, λυπάμαι που έχει φύγει. Ε, ε, ότι βγάζει το καπέλο. Ναι, νομίζω αξίζει ε, αυτό στη Ρουμανία. Για μας όλοι οι φάκελοι ήταν ίση σημασίας. Ε, σε ό,τι φορά την Γκρέκο, αναλύουμε κάθε σημείο της Γκρέκο, αλλά θα πρέπει να δει και το Βέλγιο, τη χώρα του. Είναι 15 συστάσεις, ε, από τις οποίες έχει υλοποιήσει μόνο μία. Θα πρέπει να αφήσουμε να μην παρέμβουμε εμείς στο έργο της Γκρέκο και να παρεμβαίνουν οι ίδιοι οι δικαστές, αν πραγματικά θέλουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πρέπει οι δικαστές να βρουν την συνένεση και να μην τα υλοποιήσουμε αυτά εμείς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, όλους όσοι πίστεψαν σε μας, γιατί η δική σας εμπιστοσύνη δεν ήταν απλά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Ρουμανίας, όχι μόνο στους εμπειρογνώμονές μας, στους διπλωμάτες μας. Ήταν ε, η εμπιστοσύνη σε μια ολόκληρη χώρα που κατήχε για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια χώρα που έδωσε τις πρώτες εξετάσεις της ε, σε αυτό το θέμα και που εγώ θεωρώ και έχω δει και πολύ ε, συμμερίζεστε την άποψή μου ε, πέρασε με πολύ καλούς βαθμούς. Σας ευχαριστώ για την εμπλοκή σας, την στήριξή σας, τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Εύχομαι και πάλι επιτυχία στο νέο κοινοβούλιο και ε, ελπίζω να έχετε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα, το πολύ σημαντικό, στο οποίο ε, ήμουν δραστήρια για 9 χρόνια, να έχετε επιτυχία, διότι η δική σας επιτυχία είναι και επιτυχία ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σας ευχαριστώ. Ε, εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, την ε, Πρωθυπουργό κυρία Νταντσίλα, τον ε, Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτ, συγχαρητήρια για την δέσμευσή σας. Αύριο θα ξεκινήσουμε μια νέα, ένα νέο εξάμεινο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναρχίσουμε στις 6, στις 18.